και θα ήθελα να ζητήσω ένα λεπτό σιγής. Ε, Ευχαριστώ. Θα τηρήσουμε τώρα ενός λεπτού σιγής. Thank you. Koleżanki i koledzy, pod oświadczeniem pisemnym... Υπάρχει γραπτή δήλωση υπαριθμών 3 με ημερομηνία Κορίνε Λεπάς ε, φετινή όπου αναφέρεται ότι η πρωτοβουλία Let's Do It έχει υπογραφεί από πλειοψηφία των συναδέλφων και επομένως σύμφωνα με το άρθρο 123 του κανονισμού θα δημοσιευτεί στα έγγραφα της Ολομελίας μας μαζί με τις υπογραφές. Μήπως κανείς θέλει να σχολιάσει. Ορίστε. Eh, η κυρία Σίζηλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστώ πρώτα για την υποστήριξή σας με τη δήλωση αυτή για το έτος των εθελοντών που δείξαμε ότι για μας έχει σημασία το καθαρό περιβάλλον. Παρακαλώ μην μείνετε μονάχα στην υπογραφή του χρόνου το 2012 η δράση αυτή του καθαρισμού του περιβάλλοντός μας θα συνεχιστεί σε όσο το δυνατόν περισσότερες πόλεις και με τον τρόπο αυτό θα υποστηρίξουν την προσπάθεια και οι διάφορες περιβαλλοντικές οργανώσεις. Yes, please, colleague. The floor is yours. Έχετε το λόγο. Now it works, yeah? Α, τώρα λειτουργεί. Σύντομα παρακαλώ. Δεν φταίω εγώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ όλες και όλους που υποστηρίζουν την πρωτοβουλία αυτή. Εργάστηκα ευχαρίστως με τις κυρίες Σίζελη, Γκόμες, Κορίν Λεπάζ, Πρόκειται για μια πραγματική πρωτοβουλία πολιτών. Δείχνει πώς οι πολίτες μπορούν να δείξουν τον δρόμο στην Ευρώπη. Γνωρίζοντας τις αμφισβητήσεις σχετικά με τις γραπτές δηλώσεις, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τα μέλη εκείνα τα οποία θεώρησαν ότι δεν ήταν ορθή η εκστατεία μας και υπόσχομαι να μην ξαναρχίσω τέτοια ιστορία με γραπτή δήλωση στην παρούσα κοινοβουλευτική θητεία. Ελπίζω να με βοηθήσετε να τηρήσω την υπόσχεσή μου. Σας ευχαριστώ και πάλι και ελπίζω να σας ξαναδώ στην επόμενη μέρα του 2012. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία της εκθέσεως ΒΕΡ